κανόνες για τη συμμετοχή στον ορίζοντα 2020. Καταρχήν ψηφίσουμε το μπλοκ 1 με την τροπολογία 138 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Οι άλλες τροπολογίες εκπίπτουν ως εκ τούτου. Περνάμε στην ε, πρόταση Κομισιόν όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μία τροπολογία 139 στη συνέχεια υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή και το νομοθετικό ψήφισμα, ονομαστική κλίση και πάλι, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Πέρας. Δεκτό το νομοθετικό ψήφισμα. Ερχόμαστε στην έκθεση Ματίας, ατζέντα για στρατηγική καινοτομία το μπλοκ υπαριθμών 1 με την τροπολογία 85 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό, εκπίπτει το μπλοκ 2. Ψηφίζουμε την πρόταση της Κομισιόν όπως τροποποιήθηκε, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι, όλες. Πέρας ψηφοφορίας δεκτό το ψήφισμα. Έκθεση Λάμπερτς, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Καινοτομίας, μπλοκ 1 με την τροπολογία 61, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές δεκτό, εκπίπτει το μπλοκ 2, η πρόταση κομισιόν όπω τροποποιήθηκε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, το ορμοθετικό ψήφισμα με ονομαστική κλίση άρχεται, ψηφίσατε όλοι, πέρας, εγκρίθηκε. Έκθεση Κρότσμαν, ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2014-2020. Μπλοκ 1 με την τροπολογία 97 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Εκπίπτει το μπλοκ 2. Η πρόταση κομισιών όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική κλίση άρχεται η ονομαστική κλίση. Σφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση The Grass Carvalho ειδικά προγράμματα για την εφαρμογή του Horizon 2020, μπλοκ 1 με την τροπολογία 71, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, το μπλοκ 2 εκπίπτει, πρόταση κομισιών, όπως έχει τροποποιηθεί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Δεκτή. Δεκτό. Ερχόμαστε στην έκθεση Huang Γκόκ, Ευρωπαϊκές Στατιστικές, μπλοκ 1, με την τροπολογία 43, με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το μπλοκ 2 εκπίπτει. Περνάμε στην πρόταση της Κομισιόν όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση. Ο κύριος Χουαγκ ζήτησε το λόγο μετά την ψηφοφορία αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μόλις εγκρίναμε μία θέση πάρα πολύ ισχυρή για το θέμα αυτό Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο θα το λάβει από εδώ και στο εξή ε, υπόψη και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι πολύ επικοδομητική γιατί θέλουμε να φτάσουμε σε δεύτερη ανάγνωση το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χωάν Γκόγκ. Περνάμε στην έκθεση Steinrock, πρόγραμμα κοινωνικής ε, αλλαγής και καινοτομίας. Το μπλοκ 1 με την τροπολογία 179, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Εκπίπτει το μπλοκ 2. Πρόταση της Κομισιόν όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ε, γίνεται δεκτό. Έκθεση ΧΑΟΚ, το πρόγραμμα για κλιματική δράση και περιβάλλον, πρόγραμμα live, τροπολογία 85 μπλοκ 1, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, εκπίπτει το μπλοκ 2 και οι άλλες τροπολογίες. Περνάμε στην πρόταση της Κομισιόν όπως έχει τροποποιηθεί, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έχουμε τροπολογία 86, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε το ψήφισμα. Έκθεση στο Λογιάν. Πρόγραμμα δράσης για τη φορολογία. Μπλοκ 1 με την τροπολογία 39. ψηφίπερ Κατά αποχές εγκρίνεται ω εκ τούτου εκπίπτει το μπλοκ 2. Πρόταση τη Κομισιόν όπω έχει τροποποιηθεί, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκταση Μπαλτασάρε, πρόγραμμα δράσης για τα τελωνία, μπλοκ 1 με την τροπολογία 42, ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται εκπίπτει το μπλοκ 2 πρόταση της Κομισιόν όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 43 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το νομοθετικό ψήφισμα τώρα με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρασε της ψηφοφορίας Εγκρίνεται το ψήφισμα. Ερχόμαστε στην έκθεση Bowles για την ασφάλεια και επανασφάλιση, το Solvency 2, το κείμενο σα σύνολο, ψήφι υπέρ με την τροπολογία 1, κατά, απόχες, εγκρίνεται, η πρόταση Κομισιόν όπω έχει τροποποιηθεί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική κλίση, άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ερχόμαστε στο ψήφισμα σε σχέση με την ε, ατζέντα ανάπτυξης της Ντόχα. Έχουμε ένα ψήφισμα των πρασίνων Ο σύνολο ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Έχουμε το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς. Το ψήφισμα λοιπόν ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στο ψήφισμα της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου. Με πολλές τροπολογίες που απαιτούν ονομαστική κλίση, 8 ονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Φύσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Πάλι με ονομαστική κλίση άρχεται. Σφίσατε όλοι. Πέρας. Απέριπτε. Τροπολογία 10. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Σφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Άρχεται η ονομαστική κλίση. Σφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Άρχεται η ονομαστική κλίση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Και αυτή απορρίπτεται. Τροπολογία 1 Τον Πρασίνο. Υπέρ. Κατά. Αποχέως απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 14 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 15 πάλι με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 με προφορική τροποποίηση. Θέλετε να λάβετε το λόγο σχετικά. Κύριε Πίτη Κάινεν. Πείτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως συν, συντάκτη μα με τον Δόκτωρα Μορέιρα αυτή τη πρώτη. Θέλω να παρουσιάσω μια προφορική τροπολογία στην τροπολογία περιθμού 5 των Σοσιαλιστών για να διαγραφούν οι αναφορέ στου μη δασμολογικού φραγμού. Διότι κατά την άποψή μα δεν είναι πρόσφορο να αναφερθούν εδώ. Με τον τρόπο αυτό το μέσο τμήμα της τροπολογίας θα έχει την εξής μορφή. Χαιρετίζει την ε, εκ νέου ανάληψη των διαπραγματεύσεων για την ε, συμφωνία για την τεχνολογία πληροφορικής που αυξάνει και την κάλυψη και τον αριθμό χωρών μέσα στην εμβέλειά της. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Υπάρχουν αντιρρήσεις για αυτή την προφορική τροπολογία. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία με την προφορική τροποποίηση υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 4 Εντάξει, ψηφοφορία ελέγχου για τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Σβήσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται πράγματι. Τροπολογία 4. <clears throat> Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Σφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 6. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Ονομαστική κλίση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Το σύνολο της ε, πρώτα ψηφίσματος άρχεται η ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε στο σχέδιο δράση για το 2020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 Παράγραφος 34 αρχικό κείμενο σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές α... εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παράφος 43 αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά Αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ερχόμαστε στην έκθεση κόπα <clears throat> εφαρμογή της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Παράγραφος 7, πρώτο τμήμα, της, ε, με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Πάλι ονομαστική κλίση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9, τροπολογία 1, με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. <clears throat> Παράγραφος 22, αρχικό τμήμα. Πρώτο τμήμα ονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα, πάλι μονομαστική, άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 2. Συγγνώμη. Παράγραφος 24. Τροπολογία 2 των πρασίνων. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Παράφος 26 το αρχικό κείμενο με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας προφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ψήφι υπέρ. Κατά. Παρακαλώ και πάλι. Από την αρχή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Μονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. πέρα. Μα απορρίπτεται. 8 με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση και πάλι άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Δεκτό. Έκθεση Γκάλα. Τεχνολογική και βιομηχανική βάση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αμήνα μάλλον. Παράγραφος 4. Αρχικό κείμενο με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Αρχικό κείμενο. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 11. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα με ονομαστική κλίση και τα δύο. Πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 17 το αρχικό κείμενο, ονομαστική κλίση, άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 20 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 25 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. <clears throat> Παράγραφος 26 το αρχικό κείμενο με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας εγκρίθηκε. Παράγραφος 27 πάλι μονομαστική κλίση, το αρχικό κείμενο, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 28 το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 29 το αρχικό κείμενο ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 31 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 33 σε δύο τμήματα με ονομαστική κλίση και τα δύο. Πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα πάλι ονομαστική άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται επίσης. 34 σε δύο τμήματα και πάλι ονομαστική κλίση άρχεται το πρώτο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 36. Το αρχικό κείμενο μονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Πράγμα 37 σε δύο τμήματα, ονομαστική κλίση και στα δύο. Πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και δεύτερο τμήμα άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας, εγκρίθηκε. Σαράντα σε τμήματα πάλι, με ονομαστική κλίση και τα δύο πρώτα τμήμα άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 44 σε δύο τμήματα πάλι μονομασκή κλίση και τα δύο πρώτο άρχεται η ψηφοφορία. Σφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα του 44 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 46 σε δύο τμήματα πάλι και τα δύο με ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα αρχιέται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 47 το αρχικό κείμενο. Αν ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράφος 48 σε δύο τμήματα με ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγω 49 το αρχικό κείμενο ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 51. Το αρχικό κείμενο, μονομαστική κλίση, άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. 52. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. 53 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και το ψήφισμα ως σύνολο με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελευταία ψηφοφορία η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης Ευρωπαϊκής Νομισματικής και Οικονομικής Ένωσης, τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Έλεγχος για την τροπολογία 6. Ψηφοφορία επαλήθευσης άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται σας υπενθυμίσω όταν βγάζετε την κάρτα σας πριν από το τέλος της ψηφοφορίας δεν μετράει η ψηφοφορία σας. Τρία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα ψήφι υπέρ. Τρία επαλήθευση ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Με τέσσερι ψήφου διαφορά απορρίπτεται. Είχατε δίκιο. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Θα κάνουμε έλεγχο και στην 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 6, αρχικό κείμενο με ονομαστική κλίση. Συγγνώμη. Όχι, όχι, έχει εκπέσει. Τροπολογία 10, ονομαστική κλίση, άρχεται η ονομαστική κλίση. Ψηφίσατε όλοι. <clears throat> Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 12 με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο στην παράγραφο 19 υπέρ κατά απόχη. Θα το ελέγξουμε. 19 παράγραφος αρχίδη ψηφοφορία για επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 13. Τροπολογία 13. Συγγνώμη ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Εκπίπτει το αρχικό κείμενο μάλλον στην ε, παραγωγή 20 υπέρ κατά αποχές δεκτό. παράγωγος 21 το αρχικό κείμενο με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 24 το αρχικό κείμενο με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκπίπτει το αρχικό κείμενο. Πάμε στην τροπολογία 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα κάνουμε έλεγχο για την τροπολογία 5 η ψηφοφορία επαλήθευσης. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Εκπίπτει το αρχικό κείμενο. Περνάμε στην τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκπίπτει το αρχικό κείμενο. Το σύνολο του ψηφίσματος τώρα με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Έγκρινεται. Συγχαρητήρια σε όλους τους εισηγητές. Όσοι φεύγουν, τους εύχομαι καλή επιστροφή στις αιστείες σας. Και τώρα ε, η κυρία Περάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ψήφισμα δεν είναι αυτό που θα ήθελα να δω εγκεκριμένο. Παρόλα αυτά είναι η εντολή που δίνει η ολομέλειά μας στη διαπραγματευτική ομάδα για την επόμενη συνεδρίαση ΣΕΡΠΑ όσον αφορά την ε, συμπερίληψη μιας κοινωνικής διάστασης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπερές. Κύριε και κύριοι, προσπάθησα να κάνω γρήγορα τις ψηφοφορίες. Παρακαλώ και εσείς να μπορέσετε με ταχύτητα να αποχωρήσετε για να μπορέσουμε να περάσουμε στην, ε, ψήφου. Για την έκθεση Ριέρα Μαδουρέλο κύριο κύριος Λάινεν έχει το λόγο. Κύριε Λάινεν.